το κατά πόσο είναι δίκαιη η δίκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το Γουαντάναμο. Η ψηφοφορία θα γίνει αμέσως μετά το πέρας της συζήτηση και του επόμενου σημείου που αφορά την Ουκρανία και την υπόθεση της Γιούλιας Τιμοσέγκο και άλλων μελών της κυβέρνησής της. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βιγγένιν για ένα, λεπτό, για ένα μισή λεπτό. Συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες θεωρούν ότι για την Ουκρανία η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προτεραιότητα για τη χώρα και για το λαό τη που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θυσιάσει τα κεκτημένα του δικαιώματα. Η σημερινή κυβέρνηση έχει αναλάβει κάποιε πρωτοβουλίε για τη βελτίωση τη νομοθεσία και την καλύτερη καταπολέμηση τη διαφθορά. Φυσικά θα πρέπει να ενισχύσουμε και να θαρρύνουμε την κυβέρνηση στι προσπάθειέ τη. Ε, η κατάργηση της ατιμορρησίας της ΕΛΙΤ θα επιτρέψει την προσέγγιση της Ουκρανίας στις προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να δώσουμε σήμερα την εντύπωση ότι προστατεύουμε την ελίτ της προηγούμενης κυβέρνησης και ιδιαίτερα την κυρία Τιμοσέγκο. Και αν απευθύνουμε έκκληση στην κυβέρνηση να μην αναμειχθεί στη, στο έργο της δικαστικής εξουσίας, με ποιο δικαίωμα εμείς ε, παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά της Ουκρανίας. Αναφέρονται η δράση προηγούμενη κυβέρνηση ε, και η συλλογική ευθύνη. Αυτό όμω είναι το επιχείρημα του ΕΛΚ που υπό το πρόσχημα της ε, συλλογική Ευθύνη προσπαθεί να ε, συγκαλύψει ατομικέ ευθύνε. Δεν είναι αυτό το νόημα του ψηφίσματο. Εμεί θέλουμε να δώσουμε περισσότερε ευκαιρίε και να θαρρύνουμε τη συνεργασία Ουκρανία-Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσέγγιση όμως που υιοθετήθηκε από το ψήφισμα είναι υπερβολικά πολιτική και ιδεολογική, γι' αυτό και θα καταθέσουμε ξεχωριστό ψήφισμα. Ο κύριος Κόχλιτσεκ. Συγγνώμη, ε, μία μπλε κάρτα προηγουμένως. Θα ήθελα μόνο να ρωτήσω τον ε, συνάδελφο, λέει ο κύριος Πόσελτ, ε, τι νόημα έχουν διακηρύξει υπέρ ε, των ε, καθολικών δικαιωμάτων του ανθρώπου όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα να συμβαίνουν ε, στην Ουκρανία. Είναι η παλιά σοβιετική νοοτροπία που λέει ότι δεν επιτρέπεται να αναμειγνυόμαστε στο ιστορικό μιας χώρας. Ιδιαίτερα όμω στην περίπτωση ενό τόσο σοβαρού εταίρου μας όπως η Ουκρανία. Η απάντηση από τον κύριο Βικένιν. Θα ήθελα να πω ότι εγώ είπα ότι δεν δικαιούμαστε να επεμβαίνουμε στα εσωτερικά μιας χώρας, ιδιαίτερα στο έργο της δικαστικής εξουσίας μιας χώρας. Γιατί εμεί ζητούμε από την κυβέρνηση να μην εμπλέκεται στα δικαστικά ζητήματα, να αφήνει ελεύθερη και ανεξάρτητη δικαιοσύνη και απ' την άλλη εμεί θέλουμε να επέμβουμε στο έργο τη κυβέρνηση. Και εμεί θα πρέπει να απόσχουμε από οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση. Υπάρχουν χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα, κύριε Πόσελτ. Ζητάτε οικουμενική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωραία, πολύ ωραία. Θα πρέπει όμως να εφαρμόζεται σε όλους κάτι τέτοιο. Sorry, Mr. You can't have blue card at the... Κύριε Τάνοκ, δεν μπορείτε να σηκώσετε μπλε κάρτα σε απάντηση προηγούμενης μπλε κάρτας. Ο κύριος Κόλιτσεκ έχει σειρά. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν στιγμές που μερικέ φορές δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που βλέπουν τα μάτια μου και αυτά που ακούν τα αυτιά μου. Ε, κάτι τέτοιο μου συνέβη και όταν διάβασα το ψήφισμα για την ε, Ουκρανία. Ε, Φαίνεται ότι κάποιοι υπουργοί και πρωθυπουργοί έχουν το ατιμόρυτο, χαίρουν ατιμορρησία σε ορισμένες χώρες. Από τη μία πλευρά πάντως το Κοινοβούλιο ζητάει συγκεκριμένη δράση κατά της διαφθορά, διαφθοράς, αλλά ε, ταυτόχρονα όταν ε, μία ε, εκπρόσωπος ή κάποιοι εκπρόσωποι προηγούμενης κυβέρνησης ε, κατηγορούνται για διαφθορά ή για κακές πράξεις, τότε λέμε ότι θα πρέπει να προστατευτούν και να μην τιμωρηθούν. Βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, αλλά ας ξεκινήσουμε από το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας διαβάσουμε επίσης και το σύνταγμα της ε, περί ισολόγως ε, χώρας για να δούμε τι γράφει και ε, νομίζω ότι αφού καθαρίσουμε τα του, οίκου τα μας τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε κηρύγματα σε άλλες χώρες. η ΓΚΟΕ μπορεί να συμφωνήσει με ορισμένα σημεία του ψηφίσματος αλλά διαφωνεί κάθετα με ορισμένα άλλα γι' αυτό δεν θα στηρίξει το ψήφισμα. Επόμενος ο κ. Γκάλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς υπάρχουν αφορμές ε, για να ασκήσουμε σαφή κριτική κατά της πολιτικής κατάστασης στην Ουκρανία. Τα μέσα τα οποία, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται οι πολιτικώς δικαιολογημένες ε, ε, καταστάσεις και διώξεις κατά της Τιμοσέγκο και όποιος επηρεάζει ε, το δικαίωμα αυτό δράσης, ε, το συνταγματικό αυτό δικαίωμα δράσης, ε, όπως για παράδειγμα του Γιουτσέγκο και όπως για παράδειγμα από την κυρία Τιμοσέγκο, καταδεικνύει πώς η δικαιοσύνη την χάνει χρήση λόγω πολιτικών καταστάσεων. Θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι διώξεις. Ο κύριος Γιαννουκόβιτς και η συμπεριφορά του αποτελεί τεστ για τη συμπεριφορά της και για την πραγματοποίηση των, ευρωπαϊκών αξιών στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ. Eh, Έχουμε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Κόβαλτ. Την δέχεστε? Ο κύριος Κόβαλ. Ευχαριστώ. Σε πολλά πράγματα συμφωνούμε και ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την εδραίωση της δημοκρατίας ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα για μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης και επίσης πόσο σημαντική είναι η προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είστε έτοιμος να δηλώσετε ότι είστε υπέρ, ε, ε, να δηλώσετε υπέρ αυτής της ενταξιακής προοπτικής της Ουκρανίας να πείτε ότι και για την Ουκρανία είναι ανοιχτό ο δρόμο και ανοιχτέ οι πύλε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δεχόταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τέτοιου είδου διατύπωση. Ευχαριστούμε να ακούσουμε και την απάντηση. Ο δρόμος της Ουκρανίας προς την Ευρώπη σίγουρα δεν θα ε, υποστηριχθεί από μια τέτοια συμπεριφορά τη κυβέρνηση. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, η κυρία Όγιουλαν, την επόμενη President. Πρόεδρε. Δεν είμαστε εδώ σήμερα για να κρίνουμε κατά πόσο είναι ενοχή ή μη η Γιούλια Τιμοσέγκο. Αυτό το θέμα δεν είναι ε, αυτό που συζητάμε σήμερα, γιατί οι Ουκρανικές αρχές ε, δεν τήρησαν τις σωστές ε, νόμιμες αρχές και καταχράστηκαν το, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Διαμαρτυρόμαστε λοιπόν κατά της κατάστασης αυτής στην Ουκρανία με τη βοήθεια του δικαστικού συστήματος κατηγορούμενοι θα πρέπει να έχουν τα δικαιώματα που τους ε, αναγνωρίζει ο νόμος και αυτά θα πρέπει να είναι ανάλογα με τις κατηγορίες που τους απαγγέλλονται. Σκοπός του ψηφίσματος είναι να επιστήσει την προσοχή των Ουκρανικών αρχών στο κράτος δικαίου και στις παραβιάσεις του κράτους δικαίου που χωρίζουν την Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που αν συνεχιστούν στο μέλλον θα αφαιρέσουν τη χώρα αυτή από το ευρωπαϊκό της μέλλον. Ευχαριστώ. Ρωμέβα Ιρουέντα. Ευχαριστώ. Ο λόγος ε, για τον οποίο ε, ασχολούμαστε με το θέμα αυτό είναι γιατί θεωρούμε ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και στην περίπτωση της Ουκρανίας προσβλέποντας στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Οι προσπάθειες θα πρέπει αυτές να βασίζονται σε αμερόληπτες, ανεξάρτητες δικαστικές διαδικασίες. Ε, εμείς ε, θεωρούμε ότι ε, ενδεχομένως όντως μπορεί να υπάρχει υπερβολική δίωξη και υπερβολικές μανοπυρικές διώξεις κατά της κυρίας Τιμοσέγκο και μελών της κυβέρνησης της. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι όλες οι δικαστικές εισαγγελικές διαδικασίες και οι δίκες εάν προκύψουν θα πρέπει να γίνονται με πλήρη διαφάνεια θα πρέπει ε, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα δικαστικά μέσα, όποια και αν είναι αυτά, δεν δεν χρησιμοποιούνται επιλεκτικά ε, και ε, βεβαίως θα πρέπει να στηρίξουμε την μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα στο σύνολό του στην Ουκρανία, δημιουργώντας ένα υψηλού επίπεδου συμβουλευτικό σώμα στην Ουκρανία, η οποία θα βοηθήσει διάφορες μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή, συμπεριλαμβανομένου και του δικαστικού τομέα τομέα. Ξεκινώντας τώρα με του ομιλητέ των ομάδων, η κυρία Μπασέσκου από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, μέσω των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατά της ε, Γιούλια Τιμοσένκο η παρούσα κυβέρνηση ε, συνεχίζει μία σειρά μέτρων που έχει λάβει κατά των μελών της προηγούμενης κυβέρνησης. Μας προβληματίζει η χρήση των δικαστικών εξουσιών και η κατάχρηση λοιπόν εξουσίας για την επίτευξη πολιτικών ωφελών εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία έτσι ώστε ε, να γίνει η απαραίτητη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και για να μπορέσει λοιπόν η δικαιοσύνη να προχωρήσει με τρόπο δημοκρατικό, διαφανή και αμερόλεπτο. Θα πρέπει επίσης ε, μια χώρα σαν την Ουκρανία οπωσδήποτε να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνοντας υπόψη την θέση που έχει ε, λάβει η Ουκρανία στα πλαίσια της ανατολικής ε, γειτονίας ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη στη Συμφωνία Εταιρική Σχέσης και την υπογραφή της. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει η κυρία Γκέργκερ Γκέριγκερτε-Εντεμπερκ. Ευχαριστώ. Μια από τι προτεραιότητε της επερχόμενης πολωνικής είναι η ενδυνάμωση τη Ανατολική εταιρική σχέση. Η Ουκρανία ω πλησιέστερος γείτονα τη Πολωνία, είναι από του πιο σημαντικού μα εταίρου και έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί περισσότερο αυτήν την ανατολική σχέση. Συμφωνώ με την ανάγκη προσέγγιση τη Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω όμω ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να συνδυαστεί αυτή η προσέγγιση με την υιοθέτηση από τη χώρα αυτή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και τι του δημόσιου βίου. Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθώ τα σκάνδαλα της διαφθοράς και τις δίκες ε, πολιτικών, όπου οι διάφορες πλευρές ανταλλάσσουν μεταξύ τους κατηγορίες, μερικές φορές με τραγελαφικό τρόπο. Φυσικά βλέπουμε προσοχή τα συμβάντα στην Ουκρανία και τις ε, δηλώσεις που ήταν πολύ μετριοπαθείς και ισορροπημένες τις είπα τις εκπροσώπου γιατί δεν μπορούμε να αναμειγνιόμαστε εσωτερικά μιας χώρας που είναι κυρίαρχη. Στα πλαίσια όμως της μελλοντική ε, συνεργασίας με την Ουκρανία χρειαζόμαστε κάποιους μηχανισμούς που θα μπορούσε να ενισχύσει το κράτος δικαίου στη χώρα αυτή. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τη σύσταση συμβουλευτικής ομάδας για τη σύγκληση της Ουκρανικής νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή τη βοήθεια σε διάφορους τομείς όπως στην κατάρτιση δικαστών. Θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας θα πρέπει να συνδυάζεται με όρους αλλά και με βοήθεια. Και ελπίζω ότι θα είναι οι βάσεις που θα ισχύσουν και στην επόμενη Προεδρία της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ντόνσκης από τους Φιλελεύθερους και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ουκρανία είναι μια δημοκρατική χώρα. Ως εκ τούτου εκφράζουμε την ανησυχία μας ε, και το μήνυμά μας προς ε, ένα σύμμαχο και φίλο. Κανείς δεν είναι τέλειος σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά έχουμε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις ε, εύλογες αρχές της δημοκρατίας και με βάση όλες αυτές τις αρχές περιμένουμε από τις ουκρανικές αρχές να μην κάνουν κατάχρηση εξουσίας και να μην ενθαρρύνουν δίκες με πολιτικό υπόβαθρο, με για πολιτικούς σκοπούς και να εξασφαλίσουν ε, την ε, διεξαγωγή δίκαιης δίκης και όχι μιας πολιτικής ενός πολιτικού ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Γιούλια Τιμοσέγκο οι πρώην, τα πρώην μέρη της κυβέρνησης δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αυτόματα ε, ένοχοι. Όλοι είναι πολίτες ε, μία δημοκρατικής χώρας πρώτα απ' όλα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ανεφορό να υπερασπίσουμε ε, τους ε, κατηγορούμενους. Θα πρέπει απλώς να υπενθυμίσουμε στους φίλους και συμμάχους μας πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Ο κύριος Στάνοκ εκ μέρους των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Πρόεδρε, η η Ουκρανία εξακολουθεί να ε, χαρακτηρίζεται από αντιπαλότητες. Η Τιμοσέγκο και τα πρώην στελέχη της κυβέρνησή της ε, διέκονται ποινικά τώρα για πράξεις που ε, έλαβαν χώρα όταν ήταν στην εξουσία. Πολύ φοβάμαι ότι ο πρόεδρος Γιαννουκόβης προσπαθεί να εξουδετερώσει τη μοναδική σημαντική πολιτική φυσιογνωμία που μπορεί να τον αμφισβητήσει. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Πορτοκαλή Επανάσταση ήταν μια άμεση άμεση αντίδραση στην απόπειρα του Γιαννικόβιτς να κλέψει στις εκλογές του 2004 η κυρία Τιμοσέγκο απολάμβανε υποστήριξη στην Ουκρανία και συγκέντρωσε ε, πολλούς, πολλά εκατομμύρια συμπατριώτες της προς υποστήριξή της. Είναι σημαντικό ότι δεν ε, ε, απεγγείλθηκαν κατηγορίες κατά του πρώην Υπουργού Υγείας, ο οποίος έλαβε τις αποφάσεις αυτές, ο οποίος περιέργο πώς έχει λάβει και πάλι υπουργική θέση σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να μην ακολουθούμε την πολιτική χειραγόρηση του συστήματος δικαιοσύνης, όπως ο σοσιαλιστή. Πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτική αμεροληψία της εισαγγελικής αρχής ε, στην Ουκρανία. Μπορείτε να απαντήσετε κύριε Βιβιανή. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Πάσκα. Σας ευχαριστώ. Το πολιτικό σκηνικό της ε, Ουκρανίας χαρακτηρίζεται από μια κυβέρνηση η οποία ε, βρίσκει, βρίσκει τις ρίζες της ε, στο σοβιετικό πρότυπο. Ε, κυρίως οι τιμοσένκο και ε, Λούσενκο έχουν φαίνεται μεγάλη γνώση αυτής της κατάστασης. Επίσης είναι υπεύθυνη για την κρίση του φυσικού αερίου που αντιμετώπισε η Ευρώπη το 2009 και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλά κέρδισαν ε, αυτοί από την κρίση του φυσικού αερίου. Ε, η ε, εγκληματικοποίηση, η ποινικοποίηση μάλλον της πολιτικής ε, ζωής βεβαίως δεν μπορεί να μας βρίσκει σύμφωνους. Από την άλλη μεριά το ίδιο γελίο είναι να λέμε ότι κανένα μέλος της κυβέρνησης Τιμοσέγκο δεν έκανε ποτέ τίποτε κακό ή τίποτε επιλήψιμο Επομένως, εάν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε την Ουκρανία ε, να αναπτύξει μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία, θα πρέπει να σταθούμε στο πλάι της, αλλά να μην λέμε ότι κάποια από τα προεξέχοντα ε, στελέχη, των οποίων τα ονόματα ενδεχομένως γνωρίζουμε, ε, θα πρέπει να έχουν ατιμορρησία ή θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Οι ίδιες για όλους. Η κυρία Ροϊτόβα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η παρούσα κυβέρνηση προσπαθεί να βρει ε, ε, πάση θυσία παραβιάσεις της κυρίας Τιμοσέγκο και άλλων μελών της κυβέρνησής της και αυτό οπωσδήποτε δυναμητίζει το δικαστικό σύστημα της Ουκρανίας. Γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν ζήσει σε σοβιετικό καθεστώς έχουν μεγάλη ευαισθησία στον τρόπο απαξίωσης σε αυτόν τον τρόπο απαξίωση των πολιτικών αντιπάλων μέσω ε, υποτιθέμενων ποινικών ε, διώξεων. Βεβαίω θέλουμε δικαιοσύνη στην χώρα αυτή και θα ήθελα να ζητήσω ε, να ακολουθηθεί η τσεχική, το τσεχικό παράδειγμα, να δοθεί δηλαδή ασυλία σε μέλη διοκόμενα της αντιπολίτευσης στην Ουκρανία που θα ζητήσουν άσυλο σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κόβαλ. Φυσικά ε, τα πραγματικά περιστατικά είναι γνωστά και εμείς ε, τασόμαστε με, στο πλευρό των ε, δυνάμων, αυτών που έχουν πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει να αντλήσουμε και κάποια συμπεράσματα και πρώτα απ' όλα η Ουκρανική κυβέρνηση γιατί στόχο εμπέδωση του δημοκρατικού συστήματο Ουκρανία είναι ο σεβασμό των δικαιωμάτων τη αντιπολίτευση. Και αυτό θα πρέπει να το δηλώσουμε ρητά και κατηγορηματικά. Θα πρέπει όμω εξίσου ρητά και κατηγορηματικά να πούμε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτή τη στιγμή ε, δεν θα έχουμε πραγματικό εξυγχρονισμό ε, και στην Ευρώπη αν υπάρχει θέση και για την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έστω μετά από μερικά χρόνια, αν δεν, που, αν δεν μιλήσουμε ρητά για την ε, ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας, τότε θα γίνουμε συνένοχοι της, α, ε, του, της ενός κακού και συντηρητικού συστήματος στην Ανατολή. Ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Τα πράγματα είναι απλούστατα. Έχουμε και εμείς να κάνουμε κάτι στη συζήτηση. Να πούμε ρητά, οι πόρτες είναι ανοιχτές, μη φοβάστε. Ευχαριστώ το λόγο κύριος Μιγκάλσκι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτά που είπε ο κύριος Ντόνσκης και είπε ότι οι Ουκρανοί είναι φίλοι και συμμαχοί μας. Όντως, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους φίλους μας. Και θα ήθελα να θέσω και την επόμενη ερώτηση. Συμφωνώ και εγώ με τις παρατηρήσεις που έκαναν οι περισσότεροι. Ούτε κι εγώ ε, είμαι ικανοποιημένο από την ε, τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη λειτουργία τη δημοκρατίας στην Ουκρανία. Θα ήθελα όμως να σας θέσω μια ερώτηση. Τι κάνατε εσεί, τι έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι έκαναν όλοι αυτοί που από καθέδρα σήμερα στυλιτεύουν την κατάσταση για την υπόθεση Τιμοσέγκο. Εσείς τι κάνατε ώστε στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις να δοθεί ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φίλος και σύμμαχος της Ουκρανίας και ότι την περιμένουμε με ανοιχτέ αγκάλες και ότι κάποια στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δεχθεί και Ουκρανούς Ευρωβουλευτές ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η τήρηση της δημοκρατίας στην Ουκρανία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από εμά. Θα ήθελα παρακαλώ να το συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτό. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα... Ο κύριος Πόσολτα έχει μπλε κάρτα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο αν ξέρει ότι εμείς στο κοινοβούλιο αυτό με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίναμε ένα ψήφισμα και εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό, όπου ε, τονίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Αυτό όχι μόνο μία φορά, αλλά σε διάφορες περιστάσεις. Κύριε Ευρωβουλευτά, το γνωρίζω. Πρώτον και δεύτερον, σας ευχαριστώ. Αλλά θα περιοριστούμε σε κάτι τέτοιο, ερωτώ και το Κοινοβούλιο και τα κοινωνικά θεσμικά όργανα μπορούν να ασκήσουν επιρροή υπέρ των Ουκρανών που δίνουν μάχη παρόμοια μάχη με αυτή που έδωσαν οι Πολωνοί και οι Τσέχοι. Να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα προς την ε, Ουκρανία για την ε, ενταξιακή της προοπτική και μάλιστα τέτοιο μήνυμα να εκπορευθεί από τη γερμανική κυβέρνηση. Προχωράμε τώρα σε διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙ. Ο κύριος Κέλλη. Ε, Ο δρόμος για την ε, δημοκρατία είναι ένας δύσκολος δρόμος ε, και άλλοι προχωρούν σε αυτόν πιο γρήγορα από ότι κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν χώρες οι οποίες βρίσκονται στο παλαιό σοβιετικό μπλοκ και που τώρα είναι μαζί μας εδώ συνάδελφοι και αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ε, ε, για την ε, Ουκρανία, έστω και αν αναγνωρίζουμε ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδο. ανάγκη είναι να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερα και όσον αφορά την κοινωνία γενικότερα και όσον αφορά τον έλεγχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όσον αφορά επίση την ανεξάρτητη δικαστική, ανεξάρτητες δικαστικές και τέλος ε, ε, δημοκρατία η οποία δεν έχει ισχυρή αντιπολίτευση δεν μπορεί να είναι ε, πραγματική δημοκρατία. Επομένως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ουκρανία να προχωρήσει στην πλήρη οδό του εκδημοκρατισμού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Η κυρία Εσάγια. Πράγματι, η ε, τρεις ποινικέ ε, διώξεις κατά της ε, κυρίας Τιμοσέγκο, τις οποίες απήντησε λέγοντας ότι πρόκειται για πολιτικές διώξεις στην ουσία, είναι γεγονός. Πρέπει να πω ότι η κυρία Τιμοσέγκο και κάποια άλλα μέλη της κυβέρνησής της κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα. Εμείς εδώ, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, δεν είμαστε δικαστήριο να αποφασίσουμε αν είναι αθώα ή ένοχη. όμως βρισκόμαστε βρισκόμαστε εδώ για να επιστήσουμε την προσοχή ε, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Ε, θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της μη διακριτική μεταχείρισης, θα πρέπει να είναι ίδια για όλους. Ε, η Λέβη Άστον τον Μάιο ανέφερε τον προβληματισμό της κυρίως όσον αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες και τις ενδεχόμενες πολιτικές σκοπιμότητες που κρύβονται πίσω ε, από αυτές. Ε, βεβαίως ε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να είναι αμερόληπτη. Κύριε Σιλβέστρη, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιλβέστρη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Η Ουκρανία είναι ε, δημοκρατία, σύμμεχο και φίλη χώρα. Η Ουκρανία όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να μεταρρυθμίσει το δικαστικό της ε, ε, σύστημα στο οποίο ανθούν πολιτικές, πολιτικής υφής δικαστικές και ποινικέ διώξεις. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ποινικοποίηση της πολιτικής ε, ζωής ε, γιατί για πολιτικούς λόγους εξαπολύονται κατηγορίες κατά των προηγούμενων των μελών της προηγούμενης κυβέρνησης. Όλοι αυτή το σύστημα ποινικών διώξεων κατά της κυρίας Τιμοσέγκο και άλλων μελών το καταδεικνύουν. Θα πρέπει η Ουκρανία να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να σέβεται το κράτος δικαίου έτσι ακριβώς όπως ορίζει ε, και το, η Ανατολική Εταιρική Σχέση την οποία έχει υπογράψει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κόρχολα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρώην Υπουργός, ε, Πρωθυπουργός κυρία Δημοσένκο. κατηγορήθηκε για πάμπολες φορές για διαφθορά και γι' αυτό δεν μπόρεσε να επισκεφτεί και τις Βρυξέλλες την Άνοιξη. Σε περίπτωση που καταδικαστεί για τις ε, κατηγορίες αυτές θα ε, τιμωρηθεί με δεκαετή φυλάκιση. Πρόκειται για κατηγορίες οι οποίες έχουν και πολιτικό υπόβαθρο, πολιτική αιτία. Αυτές οι επιλεκτικές διώξεις ε, ε, κατά μελών της αντιπολίτευσης και η έλλειψη διαφάνειας του δικαστικού συστήματος. Τέτοια ζητήματα είναι σημαντικά για την εμβάθυνση των σχέσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της Ουκρανίας. Θα πρέπει να συνεχιστούν λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες ξεκίνησαν στην Πρωτοκαλία Επανάσταση. Ευχαριστώ και τελευταίος ομιλητής ο κ. Ματούλα. Ευχαριστώ. Το ψήφισμα για τις διώξεις, για τις υποθέσεις κατά πρώην μελών της Ουκρανικής κυβέρνησης είναι απαραίτητο γιατί θα πρέπει να σεβόμαστε τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώτα απ' όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μας ανησυχεί τόσο η κουρανική δικαιοσύνη, αλλά η πιθανότητα κρατικής παρέμβασης στο έργο της δικαιοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αρχών και αξιών και θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, τα πρώην μέλη της Ουκρανικής κυβέρνησης και να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή του τεκμηρίου της αθωότητας και το σεβασμό της, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ανθρωπίνων, Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θέλουμε μια σύγκληση της Ουκρανικής νομοθεσίας προς το κοινοτικό κεκτημένο. Η επιτυχία των Ουκρανικών μεταρρυθμίσεων θα εξαρτηθεί από την πρόθεση και το σεβασμό των δημοκρατικών αξιών, του κράτους δικαίου και της διαφάνειας. Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες της βάρος κυρίας Τιμοσέγκο και των πρώην μελών του Υπουργικού Συμβουλίου της, ε, δεν θα πρέπει ε, οι ισχυρισμοί αυτοί να αποβούν εις βάρος της δημοκρατίας, γιατί αναφέρονται κάποιες κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας. Ο Επίτροπος Έτιγκερ. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία με μεγάλη προσοχή. Όπως και εσείς ως Κοινοβούλιο και η ομάδα του Κοινοβουλίου σε συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα πρώην μέλη της κυβέρνησης της κυρίας Τιμοσένκο και γιανοσένκο Από την αρχή του έτους ε, εκφράσαμε τις αμφιβολίες μας σε σχέση με, το, με, τα, με τις αιτίε αυτών των ε, κατηγοριών και παρακολουθούμε με, από στεν, στενά την κατάσταση. Πριν από λίγες ημέρες ε, δημοσιεύθηκε και μια έκθεση προόδου για την Ουκρανία η οποία απεικονίζει την κατάσταση στη χώρα. Το ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στην χώρα καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η έκθεση τονίζει ότι η τήρηση του κράτους δικαίου στις ποινικέ ε, διώξεις και στα ποινικά μέτρα που λαμβάνονται καθώς και θα πρέπει και ότι το αμερόληπτο δικαστικό σύστημα είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά προκειμένου να μην την χάνει κατάχρηση στο ποινικό σύστημα. Σε περιπτώσει που εμπλέκονται τα μέλη της πρώην κυβέρνηση, θα πρέπει σαφώς να γίνει διάκριση μεταξύ ποινική και πολιτικής ευθύνης προκειμένου να μην υπάρχει αυθαίρετη προσέγγιση της δικαιοσύνης να μην είναι υπερβολική λήψη μέτρων σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και την επιβολή ποινών. Πολλοί πιστεύουν ότι το δικαστικό σύστημα στην Ουκρανία υπόκειται σε μεγάλες πιέσεις Ελπίζουμε στο μέλλον να τροποποιηθεί η νομοθεσία για την ε, δικαστική μεταρρύθμιση και να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης προκειμένου να, να μην υπάρξουν άλλες τέτοιες αμφιβολίες. Θα ήθελα να τονίσω ότι το κράτος δικαίου στην Ουκρανία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβει υψηλή σημασία. Πρόκειται για μια χώρα με την οποία έχουμε στενή εταιρική σχέση και οικονομική ενσωμάτωση βάσει συμβατικών σχέσεων και αυτό επιθυμούμε για το μέλλον. Η ομαλή και εύρυθμα λειτουργούσα δικαιοσύνη είναι προς αυτήν την κατεύθυνση κάτι το αναπόσπαστο. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε υπερβολικά συστήματα, αλλά θέλουμε να αλλάξει το σύστημα στην Ουκρανία προκειμένου να υπάρχει η εγγύηση της αμερόληπτης και δίκαιης ε, δίκης. Είμαστε ε, πεπισμένη ότι η σταθερότητα στην Ουκρανία και η εμπιστοσύνη των πολιτών ε, στο κρατικό σύστημα θα εξαρτηθεί από αυτές τις εξελίξεις. Όπως είπα ήδη, η ταχύτητα της προσέγγισης μας προς την Ουκρανία θα εξαρτηθούν από την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και της αρχής του κράτους δικαίου. Και για όλα αυτά θα πρέπει φυσικά να δοθούν εγγυήσεις. Δεν επιτρέπεται να τίθενται ένα αμφιβόλο αυτές οι διαπιστώσεις. Αυτά θα καθορίσουν την μελλοντική πολιτική εταιρική σχέση. Ε, στις επόμενες ε, ε, εβδομάδες θα λάβουν χώρα συνεδριάσεις της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας και θα ανακύψουν, θα εξεταστούν τέτοια σημαντικά θέματα για τις σχέσεις μας και θα αποσταλούν σαφή μηνύματα προς την Ουκρανία για τη σημασία των μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό. Και είμαστε ικανοποιημένοι από την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας να κλείσει τις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία εταιρική Σχέσης πριν τα τέλη του χρόνου. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό και να πετύχουμε και την ε, εταιρική σχέση και την οικονομική σχέση, οικονομική ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει η Ουκρανία να προωθήσει τις αναφερόμενες μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, τις εκλογές και επίσης η χώρα θα πρέπει να συνεχίσει την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν είναι μόνη της, ωστόσο, η Ουκρανία στον αγώνα αυτό. Θα πρέπει όμως να μας αποδείξει τη θέλησή της για τις μεταρρυθμίσεις αυτές και τη θέληση της να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία στις προσπάθειές της αυτές για την εξαγωγή των μεταρρυθμίσεων. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι σεβόμαστε ασφαλώς χωρίς οποιοδήποτε σχόλιο μια σωστή διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Χρειαζόμαστε τις ιστορικές αυτές μεταρρυθμίσεις ε, στην Ουκρανία προκειμένου να υπάρχει προσέγγιση και προς τις αρχές αλλά και προς την αντιπολίτευση της χώρας αυτής. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τελειώσαμε και τη συζήτηση για την Ουκρανία. Μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. The first item... Το πρώτο θέμα είναι η ψηφοφορία για έξι προτάσεις ψηφίσματος για τη Μαδαγασκάρη.